μη πολλωμένη συζήτηση εδώ. Αν θέλετε να υπάρξει δέσμευση ολόκληρη τη Ολομέλεια, Σα παρακαλώ, διακόπτη πάλι πρόεδρο. Σα παρακαλώ. Ε, Σα ευχαριστώ. Σα ανακοινώνω ότι έλαβα πρόταση ψηφίσματο μετά την ολοκλήρωση τη συζήτηση. Η ολοκλήρωση τη συζήτηση έγινε τώρα και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στι 11.30. Και τώρα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, περνάμε στις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν, εξ ονόματος του Συμβουλίου, θα δώσω το λόγο στην Υπουργό Γιώρη. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αύριο θα ψηφιστεί το ψήφισμα για την ε, διαδικασία ένταξη του Μαυροβουνίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει δέσμευση να υποστηρίξει την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει όμως να πείσουμε και την κοινή γνώμη. Το ψήφισμα που θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο δείχνει την ε, σημασία αυτής της αναγνώρισης. Το Συμβούλιο ε, συμμετέχει δραστήρια. Έχει εξασφαλίσει μια συνένεση από το Δεκέμβριο του 2010. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει να είναι υπέρ της συνέχισης της διαδικασίας Ένταξη των χωρών της Δυτικής, των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουγγρική Προεδρία επίσης συμμετέχει δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για τις προσπάθειές του. Με αυτό το ψήφισμα ε, βοηθάει ε, και επιβεβαιώνει τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου. Κάτι που βοηθάει πολύ στην ένταξή του. Πολλές φορές έχουμε τονίσει την ε, σημασία της ε, διαδικασίας που λαμβάνει η χώρα στο Μαυροβούνιο. Η σταθερότητα της χώρας στηρίζεται έχει, έχουμε, έχουμε ε, ενισχύσει τη σταθερότητα του Μαυροβουνίου με αυτόν τον τρόπο και το Μαυροβούνιο με τη σειρά του μπορεί να βοηθήσει τη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων. Σε λιγότερο από, πριν από λιγότερο από ένα χρόνο το Μαυροβούνιο κατάφερε να εξασφαλίσει την κατάρριξη των θεωρήσεων για ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η ευρωπαϊκή προοπτική αποτελεί ατμομηχανή για τις εξέλιξεις στη χώρα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ε, την, ε, τις προσπάθειες των υποένταξη χωρών. Βέβαια, πρόοδος μπορεί να γίνει πολύ ακόμα. Προκύπτουν καινούριε υποχρεώσει, καινούριε δεσμεύσει ε, και εμείς ε, έχουμε καινούριε προσδοκίες. Σχεδόν ε, καθημερινά λαμβάνουν χώρα συναντήσεις μεταξύ εμπειρογνωμόνων και συζητούνται θέματα ένταξης του Μαυροβουνίου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα δράση το οποίο επικαιροποιείται για το οποίο η Κομισιόν μάλιστα έχει προετοιμάσει την απάντησή της. Μας ε, ενδιαφέρει η μεθοδολογία, ε, δηλαδή με, με άλλα λόγια, σε αυτό το πρόγραμμα δράση του, το του Μαυροβουνίου είναι αποτέλεσμα διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία κλειδιά στα οποία πρέπει να ε, επιτευχθεί πρόοδος. Το Νοέμβριο του 2010 η Κομισιόν ανέφερε ποιες είναι οι προτεραιότητες. Σταθερότητα του κράτους δικαίου, οι πρόσθετες μεταρρυθμίσεις και η διεύρυνση των δυνατών δράσης του, των κρατικών αρχών. Και επίσης η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά όχι μόνο από νομικής πλευράς. Ε, είναι σημαντικά γιατί δείχνουν ότι η κατάσταση αλλάζει Μην ξεχνάμε επίσης ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την, ε, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Μαυροβούνιο να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα πιο αποτελεσματικά. Χρειαζόμαστε συνεργασία σε αυτό το τομέα με το Μαυροβούνιο για να συνεχιστεί η διαδικασία και για να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις το Μαυροβούνιο θα πρέπει να πετύχει προόδο σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα πρέπει να δούμε αυτά αποτελέσματα από την πλευρά του Μαυροβουνίου. Το Μαυροβούνιο είναι πολύ σημαντικό στα πλαίσια της ε, περιφερειακής συνεργασίας. Είναι γείτονά μας. Ε, προσμένουμε σε βελτίωση ακόμα περαιτέρω της συνεργασίας αυτής και πιστεύουμε ότι το Μαυροβούνιο μπορεί να μας βοηθήσει στη συνεργασία μας και με τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης ε, φιλοξενεί το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας και άλλου είδους ε, περιφερειακά φόρα. Χάρη σε αυτή την συνεργασία μπορούμε να θεωρούμε το Μαυροβούνιο θετικό, πολύ θετικό παράδειγμα. Επίσης ε, πρέπει να περιγράψουμε σωστά την τη σημερινή κατάσταση έτσι ώστε να βοηθήσουμε στις μεσολαβικές προσπάθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για, σε όλους. Ήθελα απλώ να πω προ τι αρχέ του Μαυροβονίου θα πρέπει να συνεχίσουν τι μεταρρυθμιστικέ του προσπάθειε και να προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τι προσδοκίε των ίδιων του των πολιτών. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπο Φιούλε. Madam President, honorable members, Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, είναι τιμή μου να ε, μιλήσω σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την διαδικασία ολοκλήρωσης του Μαυροβουνίου και να αρχίσω όπως ε, τελείωσε η Προεδρία συγχαίροντας ε, τον κύριο Τάνοκ που είναι ο για την ένταξη του Μαυροβουνίου ε, και όλους τους βουλευτές που συνέβαλαν στη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Το Κοινοβούλιο παίζει ρόλο κλειδί για τη διεύρυνση και νομίζω πως η συντονισμένη δράση όλων των ευρωπαϊκών θεσμών μπορεί να πετύχει περισσότερα. Το, η γενική πρόοδος του Μαυροβουνίου προς την πλήρωση των κριτηρίων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αξιοσημείωτη. Υπάρχει αυξανόμενη πολιτική συνένεση. Η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο γιατί έχει δημιουργήσει το νομικό και θεσμικό της πλαίσιο. Επίσης είναι δεσμευμένη στην περιφερειακή συνεργασία και υπάρχει ένα ε, ε, συμπαγές ρεκόρ στις, στις διαρθρωτικές ε, αλλαγές καθώς και μεγάλη πρόοδο στο οικονομικό και κοινωνικό κεκτημένο. η η ευρωμαϊκή απόδοση του καθεστώτος ε, χώρας προς ένταξη είναι ένα σημαντικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική διεύρυνση. Η χώρα έχει μπει τώρα σε μια καθοριστική φάση. Το καθεστώς υποψήφιας χώρας είναι μεγάλη ευθύνη για το Μαυροβούνιο τα απτά αποτελέσματα χρειάζονται, ούτως ώστε το Μαυροβούνιο να είναι σε θέση να κινηθεί προς την επόμενη φάση ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είμαι βέβαιος ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα στείλει το κατάλληλο μήνυμα στο Μαυροβούνιο αναγνωρίζοντας ε, τις ε, περισμένες επιτυχίες αλλά και τις σημαντικές προσδοκίες πως η μεταρρυθμιστική διαδικασία θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα και ότι όλες οι προκλήσεις κλειδιά στο δρόμο του Μαυροβουνίου προς την ένταξη στην Ένωση θα αντιμετωπιστούν ε, καταλήλως. Εγώ συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου, τον κύριο Λούτσιτς, την περασμένη εβδομάδα ε, με διαβεβαίωση για την ε, αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις και τις προτεραιότητες κλειδιά κατά την άποψη της Κομισιόν. Τον Φεβρουάριο μετά από δημόσια διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και συνομιλίες με τις υπηρεσίες της Επιτροπής η κυβέρνηση υιοθέτησε ένα πρόγραμμα δράσης ώστε να αντιμετωπίσει αυτές τις προτεραιότητες. Είναι τώρα πολύ σημαντικό να εστιαστεί αυτή στην εφαρμογή και να φτιάξει ένα σωστό, μια σωστή ε, πορεία. Οι βασικές προτεραιότητες που εκτίθεται σε δική μας ε, γνωμοδότηση είναι μια σημαντική αλλά ε, ε απτή πρόκληση που απαιτεί την δέσμευση και την προσήλωση όλων των αρμόδιων φορέων στο Μαυροβούνιο. Ε, Παλιότερα είπαμε ποια είναι η σημασία της αντιμετώπισης των θεμάτων κλειδιών, καθώς και το κεφάλαιο 23 νωρίς στην προταξική διαδικασία. Η... Τα επιτεύγματα σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτικοποίηση της δημόσιας διοίκησης την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος καθώς και την αποτελεσματική δράση αγώνα κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος πράγματα που αργότερα θα εξασφαλίσουν τις ομαλές διαπραγματεύσεις και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο θα πρέπει να βελτιώσει και το εκλογικό πλαίσιο σε συμφωνία με τη σύσταση του ε, ΟΣΑ και, ε, της ΟΑΣΕ και της Επιτροπής της Βενετίας. Χρειάζεται ενίσχυση του Κοινοβουλίου, μια σημαντική προτεραιότητα της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου, η πραγματική συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι δε απαραίτητη, ιδιαίτερα όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών. Περαιτέρω προσπάθειες χρειάζονται για την ενίσχυση της πολιτικής κατά των διακρίσεων και συγκεκριμένα την ισότητα των φύλων αλλά και την πραγματική προστασία των ευάλωτων ομάδων. Βιώσιμες λύσεις χρειάζονται εξάλλου για τους εκτοπισμένους. Άλλα προβλήματα που εντοπίζονται στην γνωμοδότηση και στο δικό σας διοψηφίσματος ε, θα πρέπει εξίσου να αντιμετωπιστούν. Το Μαυροβούνιο χρειάζεται να ενισχύσει τις διοικητικές του ικανότητες καθώς και να αναβαθμίσει την προετοιμασία του σε διάφορους τομείς του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Το μέλλον του Μαυροβουνίου αναμφίβολα ε, βρίσκεται εντός της Ένωσης και θα πρέπει υπεύθυνα να ενεργήσουμε η αξιοπιστία της πολιτικής διεύρυνσής μας βασίζεται στις χώρες, στη σεβασμό των χωρών διεύρυνσης, των όρων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον σεβασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι στις ε, προσένταξη χώρες. Είναι προς το συμφέρον όλων να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε επιτέγματα και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Η απόδοση του Μαυροβουνίου φέτος θα αξιολογηθεί στο πακέτο διεύρυνσης που θα εκπονηθεί για τον Οκτώβριο του 2011. Η Κομισιόν ε, θα πρέπει να αξιολογήσει αν το Μαυροβούνιο έχει επιτύχει τον απαραίτητο βαθμό συμμόρφωση προς τα κριτήρια ένταξης και συγκεκριμένα τις 7 προτεραιότητε κλειδιά που εκτίθενται στην ε, γνωμοδότηση. Θα είναι σε θέση να συστήσει την έναρξη των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων μόνο τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα το λόγο έχουν ε, οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων ξεκινώντας από το ΕΛΚΑ ο κύριος ε, Τάνοκ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε Επίτροπε επισκέφθηκα την περιοχή προσφάτως με τον σκιώδη συγητή για να δούμε ποια είναι η χώρα η οποία ήταν η πρώτη που επέτυχε το καθεστώς της υποψηφίου χώρας. Είδα ότι μία κυβέρνηση μπορεί να λειτουργήσει σωστά αν, ακόμη και είναι πολύ μικρή. Ο κύριος Ζουκάνοβιτς και ε, ο κύριος Λούκτσεκ ε, ήταν ρεαλιστές και γι' αυτό προσέγγισαν σωστά το θέμα για να επιτύχουν την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα βέβαια θα πρέπει το Μαυροβούνιο να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις προσδοκίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως Έχω ε, δει ε, την έκθεση, συμφωνώ σχετικά με την διαφθορά και θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα με τα οποία να μετρήσουμε την πρόοδό τους διότι ε, θα χρειαστεί ένα πρόγραμμα δράσεως για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Βλέπουμε ότι η χώρα αυτή ξεκινά τώρα τις διαπραγματεύσεις σαν επίσημος υποψήφιος για προσχώρηση και και απορώ πώς επιτρέπεται αυτό και ε, γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις ε, διότι από, διαβάζοντας συνθήκες δεν βλέπω πώς αιτιολογείται. Επίσης ε, στην Ποντγκορίτσα και σε άλλες περιοχές όπου προσπαθούν να επιτύχουν καθεστώς υποψηφιότητος θα υπάρξει απογοήτευση και γι' αυτό ελπίζω ότι εάν ενισχύσουμε το Μαυροβούνιο δεν θα μειώσουμε το ενδιαφέρον τους για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση γιατί θα πρέπει να αποτιμήσουμε μόνο τα αποτελέσματα και όχι την κατάσταση των γειτονικών χωρών στα Δυτικά ε, Βαλκάνια. Είναι μία μικρή χώρα με ανάπτυξη και σταθερή οικονομία από όταν ε, από την Σερβία. Έχει μία ε, η διαφορά με ε, την Κροατία που θα επιληθεί ειρηνικά στο ε, δικαστήριο και χωρίς να είναι μέρος της Ευρωζώνης έχει μία οικονομία η οποία βασίζεται στον τουρισμό και εις ε, ε, ε, χιτήριο αλουμινίου. Γενικώ είναι μια εξαιρετική οικονομική κατάσταση και θαυμάσια νέα για την κατάσταση των Δυτικών Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Εξ ονόματος του ΕΛΚ τώρα ο κύριο Ιμπριζάντζικ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως σκιώδηση συγκεκριά εκ μέρου του ΕΛΚ ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τάνοκ για την πολύ καλή συνεργασία και την εξαίρετη εκθεσή του. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να στηρίξουν αυτή την έκθεση αύριο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Τον περασμένο Δεκέμβριο το Συμβούλιο των Υπουργών έδωσε στο Μαυροβούνιο ε, το παραχώρηση το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα. Αλλά το Μαυροβούνιο αυτό που βέβαια που στοχεύει είναι η πλήρης ένταξη. Από την ανεξαρτησία του και μετά έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο. Σήμερα η εκπρόσωπος του Συμβουλίου μας είπε ότι το Κοινοβούλιο θεωρείται ε, επιτυχία ε, ε, το έργο του, Κοινοβουλίου θεωρείται, ε, του Μαυροβουνίου θεωρείται επιτυχές. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις. Η Κομισιόν θα πρέπει να καθορίσει το συντομότερο δυνατό μια ημερομηνία για την ένταξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν ιδιαίτερα στο δικαστικό τομέα και να καταπολεμηθούν συγκρούσει συμφερόντων στον κρατικό τομέα. Οι προτεραιότητες που θέτει η Κομισιόν σίγουρα θα πρέπει να καταστούν προτεραιότητες και των αρχών του Μαυροβουνίου. Όμως ήδη έχουν προβεί σε πολύ θετικέ μεταρρυθμίσεις και αυτό είναι ευχάριστο. Ο πρέσβης του Μαυροβουνίου είναι παρόν και ε, περιμένουμε ανυπομονησία τη μέρα που θα καλωσορίζουμε όχι μόνο τον πρέσβη του Μαυροβουνίου, αλλά και τους ευρωβουλευτές του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Φάρμ, για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ συνάδελφοι και ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ για την πολύ επικοδομητική συνεργασία. Είμαστε ευτυχείς που το Μαυροβούνιο έχει ξεκινήσει την πορεία του προς την Ένωση και η Κομισιόν πρέπει να ξεκινήσει την ενταξιακή ε, διαδικασία όσο γίνεται πιο σύντομα. Ε, βεβαίως το Μαυροβούνιο θα πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της Ένωσης, αλλά το καθεστώς υποψήφιας χώρας είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη ώστε να εξασφαλίσει ότι ολόκληρη η πρώην Ιουκοσλαβία θα έχει μέλλον στην ε, Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μαυροβούνιο θα μπορούσε να δώσει το παράδειγμα και για τις υπόλοιπες χώρες και είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός για ολόκληρη την ε, περιοχή και τη σταθερότητα της. Ε, το Μαυροβούνιο είναι μια μικρή χώρα που είναι πολύ ε, δεσμευμένη στην περιφερειακή συνεργασία, έχει καλές σχέσεις με όλους τους, όλους τους γείτονες. Υπάρχουν ωστόσο κάποιοι τομείς όπου χρειάζονται βασικές μεταρρυθμίσεις όπως το δικαστικό σύστημα, η μετακίνηση προς ένα αυτό καθ' αυτό κράτος δικαίου, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα. Το δικαστικό σύστημα χρειάζεται μεγαλύτερη όθηση, μεγαλύτερη στήριξη για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι απαιτήσει τη Ένωση. Θα πρέπει επίση να εξασφαλίσουμε ότι το Μαυροφόνιο θα βελτιώσει τη θέση των γυναικών, θα εξασφαλίσει την ελευθεροτυπία και τα βασικά δικαιώματα των εργαζόμενων, των μειονοτήτων, καθώ και να αναπτύξει την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να ξεχνάμε πω όλοι αυτοί οι παράγοντε είναι καθοριστική σημασία για τι επερχόμενε ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Θα ήθελα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσουμε το Μαυροβούνιο όσο γίνεται πιο σύντομα στην Ένωση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Εξ ονόματο τη Άλντο, ο κύριο Βάγκελ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Τάνοκ για την έκθεσή του και για τη συνεργασία στην κατάρτισή του. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, προσπάθεια να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στο Μαυροβούνιο κατά τρόπον ώστε η χώρα να μπορέσει να γίνει μέλος θα πρέπει αυτό να δοθεί σαν δυνατότητα και σε όλες τις άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων διότι για το Μαυροβούνιο ήταν βασικό να γίνει υποψήφια χώρα αλλά τώρα πρέπει να ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση του Μαυροβουνίου πρέπει να επιτύχει πολλά. Πρέπει να αναβαθμίσει την διοίκησή της, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και ε, να έχει περισσότερες ε, δικαστικές αποφάσεις να επιδείξει σε μία μέρα όμως σαν σήμερα εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει προστασία όλων των μειονοτήτων και ότι οι αρχές αυτές θα εφαρμόζονται. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις επίσης πρέπει να έχουν μία καλύτερη θέση στην κοινωνία και ελπίζω κύριε Επίτροπε ε, ότι θα μπορέσουμε όπως μου είπαν στο Μαυροβούνιο όταν το επισκεφθήκαμε ότι οι σχέσεις με τη χώρα αυτή θα μπορέσουν να αναπτυχθούν χωρίς να εμπλακεί η Σερβία. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο έχουμε διδαχθεί από το παρελθόν, δεν πρέπει να το επαναλάβουμε διότι είναι βλαβερό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, κυρία Λούνατσεκ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να ευχαριστήσω τον Charles Τάνοκ. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σορπμένη και εξαιρετική συμφωνούμε ότι ε, λυπούμαστε για την, διαχωρισμό της έναρξη των διαπραγματεύσεων από την χορήγηση του Καθεστώτο ε, υποψηφίας χώρας. Ε, και εγώ θέλω να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Και χαίρομαι που ακούω από την Ουγγρική Προεδρία που επίσης υποστηρίζει την διαδικασία διεύρυνση. Ελπίζω ότι ε, θα παρουσιαστεί πρόοδος φέτος, το αργότερο ε, μετά την έκθεση πρόοδου. Ε, το Μαυροβούνιο έχει κάνει πρόοδο, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, στην καταπολέμηση των διακρίσεων και στην καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος ζητούμε από τις κρατικές αρχές να αποφύγουν την ε, πίεση στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που ε, ερευνούν θέματα που έχουν σχέση με το οργανωμένο κλίμα και την διαφθορά. Θα πρέπει να τις υποστηρίξουν, να τις βοηθήσουν να υποστηρίξουν το κράτος της, κοινωνίας, της οργανώσης κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει να έχουν φωνή και να μπορούν να δράσουν. Το άλλο θέμα είναι η κατανόηση των διακρίσεων. Υπάρχουν πολλέ ακόμα ομάδε του πληθυσμού ε, οι οποίε υφίστανται διακρίσει παρόλη την ομοθεσία Ε, γυναίκες, ε, ισότητα των δύο φύλων και η Ρωμά, για παράδειγμα. Τέλος, ε, το Μαυροβούνιο Σύνταγμά του ορίζεται ως οικολογικό κράτος. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια πολύ όμορφη φύση, ακτή και βουνά, αλλά ε, θα πρέπει να προστατευτούν και αυτή τη ε, στιγμή δεν γίνονται επαρκείς μελέτες περιβαλλοντικής προστασίας και χωρίς ε, αυτές η φύση κινδυνεύει να καταστραφεί. Ελπίζω ότι η χώρα αυτή θα προχωρήσει και σε αυτό το τομέα με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών και με τη χρήση διαφανών διαδικασιών σε φυσικού κάλους περιοχές. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τους υπόλοιπους εγγεγραμμένου ομιλητές. Σας παρακαλώ ωστόσο να σέβεστε το χρόνο ομιλίας σας. Το λόγο έχει ο κύριος Σόφλιν για 1,5 λεπτό. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε ε, συμφωνώ με όσα ελέγχθησαν μέχρι τώρα ότι το Μαυροβούνιο έχει κάνει σημαντικές πρόοδους για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που ξεκίνησε άσχημα. Χρειάστηκε ε, να, ε, να αντιμετωπίσει την κατάρρευση του κομμουνισμού και του κράτους και να δημιουργήσει κάτι καινούριο πάνω στα ερήπια του παρελθόντος. Πράγμα που δεν είναι εύκολο διότι ορισμένοι ορισμένοι παραμένουν έχοντας απλώς αλλάξει μορφή. Χρειάζεται όμως ένα ευρωπαϊκό μέλλον το οποίο δεν επέτυχε λόγω της αποτυχημένης ενώσεως με την Σερβία. Υπάρχουν βέβαια τα δεινά που επακολούθησαν το σοβιετικό παρελθόν, η διαφθορά, η εγκληματικότητα και η ε, ε, διεργασίες ή στη διοίκηση και στη δικαιοσύνη θα χρειαστούν βελτίωση και πρέπει να προετοιμαστούν για να μπορέσουν οι αποδέκτες του επομένου συστήματος να υποφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχει ε, εκπαιδευτεί η κοινή γνώμη και να μπορέσει να παρακολουθήσει ικανοποιητικά για να επιτύχει την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Το λόγο η κυρία Βλασίκοβα Πενόβα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόοδος στην διαδικασία ολοκλήρωσης ε, θα βοηθήσει το Μαυροβούνιο η χώρα ήδη είχε εξασφαλίσει σημαντικό βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας ενώ έχει σημειώσει πρόοδο και σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των κριτηρίων της ε, Κοπενχάγης αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, τη μεταρρύθμιση ε, του δικαστικού σώματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης χρειάζονται πρόοδοι στην μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και στην ενίσχυση του ρόλου του Εθνικού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται επίσης ε, καλύτερη προσπάθεια στην ε, διασφάλιση της ελευθερίας του τύπου, για το μέσο μαζική ενημέρωση, την μείωση των διακρίσεων, την προστασία των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και των Ρωμά, στην ε, περιφερειακή συνεργασία και στις ε, καλές σχέσει γειτονία, ε, που είναι προαπαιτούμενο για μια επιτυχή διαδικασία ένταξη. Το Μαυροβούνιο έχει πολύ δρόμο λοιπόν μπροστά του για να ικανοποιήσει τα κριτήρια και να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα Πρέπει να του δοθεί όμως η χώρα, ε, το καθεστώς της ε, υποένταξης χώρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κούκαν για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρία Υπουργέ, ε, συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ειλικρινά τον εισηγητή κύριο Τάνοκ για την εξαιρετική του έκθεση και την πολύ καλή προετοιμασία του ψηφίσματος. Το Μαυροβούνιο έχει σημειώσει καλή πρόοδο στην ενταξιακή διαδικασία. Η χώρα παίζει επίσης επικοδομητικό ρόλο στη διατήρηση της περιφερειακής ε, σταθερότητας. Είναι σε μια καλή πορεία, πράγμα που επιβεβαιώθηκε πέρυσι από την Συμβούλιο και την Επιτροπή που χορήγησαν στο Μαυροβούνιο το καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ε, ε, είμαι βέβαιο ότι τα υπόλοιπα κριτήρια για την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα, θα, θα, πληρωθούν σύντομα ώστε να ξεκινήσουν οι ταξικέ διαπραγματεύσει. Μέχρι ότου συμβεί αυτό, το, η κυβέρνηση του Μαυροβούνιου Μαυροβουνίου χρειάζεται να εστιάσει την προσοχή σε πρόοδο για τις ε, τομείς κλειδιά που έχουν σαφώς αναφερθεί. Θα τις απαριθμίσω σύντομα. Κράτος δικαίου, καταπολέμηση διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, εκλογική νομοθεσία, ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Κοινοβουλίου απέναντι στην κυβέρνηση και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος καθώς και της εισαγγελία είναι σημαντική. Η διαφθορά που υποβαθμίζει τους θεσμούς και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης η... Τέλος, είμαι ικανοποιημένο που βλέπω ότι το Μαυροβούνιο διαρκώς προχωρά στην, στην διαδικασία ολοκλήρωσης και ελπίζω πως το Συμβούλιο θα αποφασίσει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τη χώρα σύντομα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο κύριος Τάλερ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, Επίτροπε Φίλε, εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τον εισηγητή Τάνοκ για ένα μέγα επίτευγμα που αποτελεί αυτό το ψήφισμα για το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι μια μεγάλη ελπίδα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων. Η χώρα δεν έχει μεγάλες δυσκολίες ε, που να την εμποδίζουν να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να γίνει πλήρες μέλος. Οι γειτονικές χώρες είναι και αυτές μελλοντικοί υποψήφοι που πιθανότατα θα βρουν στο Μαυροβούνιο ένα παράδειγμα προς μίμηση. Εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση του κ. Λούξη, αλλά και να τονίσουμε προς, αυτού, την ίδια κυβέρνηση ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών, να το πούμε πως ε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμα και όταν επικρίνουν δεν είναι εχθροί τους, αλλά κάτι που θα, μας βοηθήσει, θα τους βοηθήσει να ενταχθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το Μαυροβούνιο λέει ότι είναι μια μικρή αλλά τίμια χώρα και ας ε, το δείξουμε αυτό σε όλους στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Μπασέσκου για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια θα εδρεωθεί ακόμα περισσότερο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δώσει το στάτους της ε, ε, ξεκινήσει μάλλον τις ενεξιακές διαπραγματεύσεις με το Μαυροβούνιο. Θα πρέπει όμως ε, το Μαυροβούνιο να ε, ικανοποιεί όλες, τα, όλες τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς ακόμα υστερεί σε σημαντικούς τομείς. Για παράδειγμα η Κομισιόν υπογραμμίζει το γεγονός ότι έχει χειροτερεύσει το φαινόμενο της ε, διαφθοράς. Χρειάζονται λοιπόν ιδιαίτερες δομές για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Από την άλλη μεριά τα δικαιώματα των μειονοτήτων και ιδιαίτερα το Ρωμά δεν ε, περιλαμβάνονται ρητά σε ένα νόμο προστασίας. Το καθεστώς αυτών των μειονοτήτων ε, δεν περιλαμβάνεται στο Σύνταγμα για παράδειγμα. Κάτι τέτοιο, μια τέτοια συμπερίληψη θα ήταν πολύ θετική. Το Μαυροβούνιο επίσης θέλει να προωθήσει την οικολογία και ένας από τους βασικούς στόχου της Ευρωπαϊκή Ένωσης είναι ακριβώς η προστασία του περιβάλλοντος. Υπ' αυτή την έννοια θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο μαζικός τουρισμός ε, μπορεί ε, να, έχει αρνητικές συνέπειες και στην ενταξιακή πορεία του Μαυροβουνίου. Επίσης, η ευρωπαϊκή προοπτική που δίδεται στο Μαυροβούνιο βοηθάει στο, η Ευρώπη να συμφιλειωθεί με το ίδιο στο παρελθόν στην περιοχή των Βαλκανίων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ταμπάζη για, Ταμπατζή, ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ <clears throat> κύριε Υφυπουργέ κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερο γιατί η Ουγγρική Προεδρία ε, θεωρεί ότι είναι προτεραιότητα να υπάρξει διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν τελικά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Οι συνάδελφοι ήδη ανέφεραν ότι ε, ε, για την προσχώρηση χρειάζεται καταρχήν να καταπολεμήσει κανείς ε, τη διαφθορά. Αλλά πέραν αυτού πρέπει να δούμε πώς προχωρούν και οι σχέσεις γυτνιάσεως. Πράγμα στο οποίο επέτυχε το Μαυροβούνιο με την Κροατία έχει υπογράψει μία συμφωνία συνεργασίας και όσον αφορά την αντιμετώπιση των μειονοτήτων το Μαυροβούνιο μπόρεσε ε, να ε, αντιγράψει το σύστημα αυτοδιοικήσεως των μειονοτήτων της Ουγγαρίας και ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσει να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 7 εγγεγραμμένους και θα μιλήσουν όλοι, αλλά σε ένα λεπτό θα τους ε, παίρνω το λόγο. Και πρώτα το λόγο έχει ο κύριος Κοτσουλόφσκι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ το Μαυροβούνιο το οποίο επέτυχε το καθεστώς υποψηφίου χώρας και ιδίως διότι ε, προχωρούν, προχωράει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο που η ιστορία της χώρας δεν είναι πολύ μακροχρόνια και ακριβώς ε, ε, χαρακτηρίζεσαι από την διαδικασία της Λισαβόνας και της Μπολόνια αλλά συγχρόνως βλέπουμε ότι υπάρχει ανεργία και μία διαφορά μεταξύ των διαθεσίμων ικανοτήτων και των αναγκών της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν όλες οι δυνατές προσπάθειες για να ικανοποιηθούν όλες οι, οι, της ε, ε, κοινωνίας και όλοι να αυξήσουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ζέμκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση αποδεικνύει καθαρά ότι το Μαυροβούνιο προσαρμόζεται όλο και περισσότερο τα στάνταρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Μαυροβούνιο σαφέστατα, αλλά να υπογραμμίσω ότι αυτή η διαδικασία έχει δύο συμπληρωματικές διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι η ευρωπαϊκή διάσταση. Οι αρχές και οι αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δείχνουν ακόμα να έλκουν τις χώρες Ευρώπης. Η δεύτερη διάσταση είναι η βαλκανική διάσταση, διότι στα Βαλκάνια υπάρχουν και άλλες χώρες τις, ε, οι οποίες μπορούν επίσης να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Είναι ένας ε, δρόμος δύσκολος, αλλά είναι δυνατόν. Οπότε, ο Επίτροπος κ. Φίλε θα μπορούσε να μας πει ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τόγκες για ένα λεπτό. Grazie. As a citizen of Ως πολίτες της Ρουμανίας με έντονη πίστη στα ωφέλη μιας ευημερούς πολυεθνικής κοινωνίας που βασίζεται στην ειρηνική συνύπαρξη και τη συμφιλίωση ανάμεσα στα έθνη, καλωσορίζω τις προσπάθειες του Μαυροβουνίου να συμμορφωθεί με τα κριτήρια της Κοπενχάγης που ταυτίζονται με τη σταθερότητα των θεσμικών οργάνων που εγγυώνται τη δημοκρατία και που αντιστοιχούν σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Το Μαυροβούνιο είναι μια κοινοβουλευτική δημοκρατία που βασίζεται σε συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά κενά στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Η διαφθορά παραμένει να είναι, μια, ε, να, είναι μια μεγάλη πραγματικότητα το οργανωμένο έγκλημα επίσης και υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Ε, ε, μάλλον κατά λάθο έσβησε το μικρόφωνο. Εγώ θα ρίνω το Μαυροβούνιο να συνεχίσει την περιφερειακή συνεργασία και να ενισχύσει τι διμερεί σχέσει με τι γειτονικέ του χώρες. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Νεβενταλόβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παρέμβαση του κ. Φίλε δείχνει ότι οι δεσμεύσει, η προσήλωση μάλλον του Μαυροβουνίου ε, στι υποχρεώσει του ε, δείχνουν το δρόμο τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται σημαντικέ κοινωνικέ αλλαγέ τα τελευταία χρόνια και στο Μαυροβούνιο και αυτό είναι πολύ θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις άλλες χώρες της ίδιας περιοχής εκτιμούμε την πρόοδο του Μαυροβούνιου και εμείς αλλά και, το, και ε, ε, ο ΟΗΕ. Σύμφωνα με το UNDP, ε, το Μαυροβούνιο μέχρι το 2015 θα πληρεί, θα έχει επιτύχει τους στόχους ηλετίας. Οι βασικές προτεραιότητες του Μαυροβουνίου είναι η ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, ε, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του. Είναι πολύ σημαντικοί στόχη και τους υποστηρίζουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπαλντασάρε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε και συνάδελφοι, δεδομένων των εξαιρετικών αποτελεσμάτων που μέχρι στιγμής έχει επιτύχει στο Τομέα της ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν ωστόσο κάποια προβλήματα όσον αφορά το κράτο δικαίου παρά τι προόδου που έχουν σημειωθεί μέσω των τροποποιήσεων ε, τη νομοθεσία για τι ποινικέ διαδικασίε και άλλε πρωτογενεί ε, νομοθεσίε, παραμένουν κάποιε σημαντικέ καθυστερήσει και αναφέρομαι κυρίως στον επίγοντα χαρακτήρα της εγγύησης, της ευθύνης και της αποτελεσματικότητας της εγγυλίας αλλά και την διαφάνεια αυτής καθώς και την ανεξαρτησία τους από τις πολιτικές παρεμβάσεις. Είναι απαραίτητες κάποιες ουσιαστικές τροποποιήσεις όσον αφορά τον διορισμό των δικαστών καθώς και των εισαγγελέων, ώστε να μην ισχύει πλέον η πρακτική σύμφωνα με την οποία ο διορισμός γίνεται μέσω της κυβέρνησης τέλος να βελτιωθεί η πρόσβαση στην δικαιοσύνη και η, να δίνεται δωρεάν νομική βοήθεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέτου. Ευχαριστώ. Η η χορήγηση του καθεστώτος της υποψήφιας ε, χώρας είναι μια πολιτική ανοιχτής ε, ε, εισόδου που έχει ασκήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Το Μαυροβούνιο βρίσκεται στην αρχή μιας πορείας που δεν θα θανούν τα ούτε εύκολη, όμως έχει αναφιλοπορίες και μπορεί να υποφεληθεί από την εμπειρία των χωρών της περιοχής που έχουν προσχωρήσει πρόσφατα στην Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή σχέση γυτνίασης και να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμβάλει αποφασιστικά στη διαδικασία συμφιλίωσης της πρώην Γιουγκοσλαβίας ε, και η ευρωπαϊκή ένταξη, ε, ολοκλήρωση όλων αυτών των πρώην χωρών της ε, Ομοσπονδίας θα θέσει τέλος σε ένα βίο παρελθόν. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έθνος του Μαυροβουνίου για το μέλλον της και για την ένταξή της ένταξή του στην Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Μίλτζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την ε, απελευθέρωση ε, του, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου θα έπρεπε να υπάρχει μια ε, πιο δημοκρατική κατάσταση αλλά είδαμε ότι υπάρχουν περισσότεροι πρόσφυγες και μια θεώρηση επισκέψεως δεν είναι ισότιμη με αυτή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό υπάρχουν υπάρχουν γραφεία τα οποία ειδικεύονται ε, στην έκδοση θεωρήσεων διαρκείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, εάν συνδυάσει κανείς το πρόβλημα αυτό με τους Ρωμά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα άτομα ε, δεν επιζητούν να παραμείνουν στο Μαυροβούνιο αλλά παρανόμως να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Μαυροβούνιο πρέπει ε, να προσπαθήσει να περιορίσει τη διαφθορά για να μπορέσει να έχει μια πιο βιώσιμη προοπτική προς την στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο Επίτροπος Φίλε. Κύριε Πρόεδρε, η συζήτησή μας ε, ήταν πολύ καρποφόρα και επιβεβαιώνει τα επόμενα απαραίτητα βήματα από πλευρά Μαυροβουνίου προκειμένου να πετύχει πρόοδο στην ένταξή του. Το σχέδιο ψηφίσματο που συζητούμε και η έκθεση τη Κομισιόν του περασμένου Νοεμβρίου αναγνωρίζουν ότι το Μαυροβούνιο έχει πετύχει πολλά, αλλά έχει επίση πολλά να κάνει στο μέλλον. Ε, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο στάδιο. Χρειαζόμαστε απτά αποτελέσματα έτσι ώστε να μπορέσει το Μοντενέγρο να περάσει, το Μαυροβούνιο να περάσει το επόμενο, στην επόμενη φάση της ένταξής του της ενταξιαστικής του διαδικασίας. Η όθηση, η ορμή που δίνει η χορήγηση του καθεστώτος υποψήφιας χώρας ε, θα πρέπει να βοηθήσει. Ε, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Ε, οι στόχοι είναι δεδομένοι. υπάρχουν προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιήσει και όταν είναι έτοιμο θα ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ο ρυθμός ε, του Κοινοβουλίου προς την ένταξή του εξαρτάται από το ίδιο το Μαυροβούνιο. Και αυτό εξηγεί ε, και τους δικούς μου δισταγμούς να σας δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ένταξη όπως μερικοί από σας μου ζητήσατε. Όμως, με την υποστήριξή μας αλλά κυρίως με την αποφασιστικότητα του ίδιου του λαού του Μαυροβουνίου, το Κοινοβούλιο μπορεί να πετύχει πραγματική πρόοδο στην ενταξιακή του πορεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε. Το λόγο έχει ο Υπουργό Γεώρη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριοι Ευρωβουλευτές, κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων διότι είναι πολύ καλό να διαπιστώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να συνεργαθεί κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να προσχωρήσει το Μαυροβούνιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας πω ότι οι ανησυχίες και τα καθήκοντα τα οποία έχουν αναφερθεί περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που έχει καταρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη διαδικασία προσχωρήσεως του Μαυροβουνίου και Βέβαια πρέπει κανείς ε, να ε, ε, σταθμίσει το χρόνο από τον οποίο η χώρα ανέλαβε το καθεστώς υποψηφίας μέχρι την αρχή των προενταξιακών συζητήσεων. Θα πρέπει εντωμεταξύ το Μαυροβούνιο να έχει εκπληρώσει 7 προϋποθέσεις, δηλαδή την ένομη η ε, καταπολέμηση της διαφθοράς και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις πρόοδους που θα έχουν επιτευχθεί και στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του έτους θα ληφθεί μία απόφαση αν μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις ή όχι. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή διότι απεδείχθη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να δώσει ένα θετικό μήνυμα στη χώρα αυτή των Δυτικών Βαλκανίων πράγμα το οποίο θα αποδεικτεί ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συνεχίζεται και υπάρχει πρόθεση προς όλες τις χώρες αυτές τις περιοχές να δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουν βέβαια κατόπιν συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Αυτό σημαίνει για τη συγκεκριμένη χώρα και ότι ενδέχεται να υπάρξουν και ε, αξιολογήσεις για την προσχώρηση της Σερβίας και της Κροατίας και οι χώρες αυτές αυτές θα πρέπει να προετοιμαστούν για να μπορέσουν διάφορες διαδικασίες να ολοκληρωθούν αν είναι δυνατόν και εντός της Ουγγρικής Προεδρίας διότι πρόκειται για γείτονες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θα πρέπει να μπορέσουν να προσχωρήσουν εφόσον έχουν επιτύχει τις προϋποθέσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ να σας ενημερώσω ότι έχω λάβει μια πρόταση ψηφίσματος για την ολοκλήρωση της συζήτησης, πέρα της συζήτησης και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30.